Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την απογευματινή μας ε, συνεδρίαση. Θα συζητήσουμε την έκθεση για το τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050. Να δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για το θέμα αυτό στη συνάδελφο Τζαβέλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές, το προσωπικό και τη γραμματεία για τη συμβολή τους στην έκθεση αυτή. Στην τελευταία ε, συνάντηση που είχαμε με τους κοιόδης ε, εισηγητές ε, συζητήσαμε τα θέματα, τέσσερα-πέντε θέματα τα οποία ήταν και αυτά τα ε, υποσυζήτηση θέματα στο επίπεδο των εισηγητών. Ε, οι πρώτες δέκα παράγραφοι είχαν διάφορα θέματα προς αρκετά δύσκολα. Ε, φτάσαμε μέχρι τις δέκα παραγράφους με τους κοιόδης εισηγητές, οπότε θα ήθελα κάποια στιγμή, αν μπορούσαμε να ενημερώσουμε και για την, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της έκθεσης. Ε, Επικεντρώνουμε στα σημεία τα οποία ήταν σημεία τριβής ή συμφωνίας ε, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Το πρώτο σημείο ήταν το θέμα των στόχων. Στην παράγραφο 3, αν δεν απατώμε, στην παράγραφο 3 υπάρχει το κείμενο. Καταλήξαμε λοιπόν ότι πράγματι υπάρχουν τρεις στόχοι της Επιτροπής για τα, τις ανανεώσιμες πηγές, την ενεργειακή απόδοση, τις υποδομές. Τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Καταλήγουμε όμως ένα κείμενο που δίνει την δυνατότητα και σε άλλες τεχνολογίες οι οποίες ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθούν ή θα εφευρεθούν στο χρονικό ορίζοντα στον οποίο, για τον οποίο συζητάμε στην έκθεση αυτή. Ένα άλλο σημείο και εκεί έχουμε μία, πρέπει να βρούμε τον ε, τρόπο της διατύπωσης στην παράγραφο 3 που μας καλύπτει όλους. Δηλαδή, ναι μεν δεχόμαστε τους τρεις στόχους της Επιτροπής, αλλά δεν είναι η μοναδική. Και νομίζω ότι σας στείλαμε τη διατύπωση και θα πρέπει να δούμε αν αποδεχόμαστε τη διατύπωση αυτή που μας βρίσκει λίγο ή πολύ σύμφωνος. Ένα άλλο σημείο ήταν ότι από τα σενάρια που εξετάζει η Επιτροπή δεν υπάρχει το σενάριο της υψηλής αποδοτικότητας σε συνδυασμό με την ε, υψηλή χρήση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή να αξιολογήσει και αυτό το σενάριο. Ένα άλλο σημείο είναι αν θα πρέπει η έκθεση να προσανατολίζεται θετικά τουλάχιστον προς ένα σενάριο. Η πρότασή μου εδώ είναι απορριπτική γιατί έχουμε τέσσερις δεκαετίες μπροστά μας για αυτή την έκθεση που συζητάμε για την υλοποίησή της. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα σενάριο, να δώσουμε μία κατεύθυνση σε ένα σενάριο γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να βρεθεί στην ενέργεια. Μπορεί η γεωθερμία, μπορεί το shale gas, μπορεί όλα αυτά να αποτελέσουν μια άλλη πηγή ενέργειας η οποία ομαλά και με πολύ υψηλή αποδοτικότητα θα μπορέσει να μας οδηγήσει στην ενεργειακή ανεξαρτησία. Τέταρτο σημείο. Κυρίες και κύριοι, οδεύουμε σε ένα μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης των κρατών μελών. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε τους μηχανισμούς συνεργασίας που ήδη υπάρχουν ή προβλέπονται από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή μηχανισμούς άλλα δίκτυα για τις διασυνδέσεις με νέες πηγές ενέργειας οι οποίες μπορούν να βρεθούν ή να υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη. Οι μηχανισμοί αυτοί, τα δίκτυα αυτά, θα συνδέουν τον Νότο με την Κεντρική Ευρώπη ή την Κεντρική Ευρώπη προς Δύση και Ανατολή. Συζητήσαμε επίσης, εφόσον υιοθετούμε το μοντέλο ενεργειακής αλληλεξάρτησης, ότι θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ένα European Support Sim for ΡΕΣ. Κάτι το οποίο είδα ότι προβλέπεται και σε μία παράγραφο από την ε, ε αναφορά του κυρίου Ρόλ, την έκθεση του κυρίου Ρόλ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εφόσον μιλάμε λοιπόν για μοντέλο αλληλεξάρτησης, δεν μπορεί να μην έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα υποστήριξης σε αυτό. Με την έκθεση δίνουμε ένα δυνατό μήνυμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το 2014 για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Και ζητάμε επίσης τη διευκρίνηση του ρόλου του ACER. Περιληπτικά αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν εξέλαβα να έχω μια καλή εικόνα των ε, τόσο όλων των ε, τροπολογιών. Αν σας έδωσα μια καλή συνθετική εικόνα ε, των τροπολογιών όσο και των συζητήσεων που είχαμε τους σκιώδεις συζητητές. Αλλά πιστεύω ότι τα σημεία στα οποία αναφέρθηκα ήταν τα επίμαχα σημεία όπου διαφωνούμε ή συμφωνούμε. η τελευταία συνάντηση, επαναλαμβάνω, έδειξε ότι μπορούμε να βρούμε ένα, τρό, ένα modus vivendi και modus οπεράντιμο περισσότερο απ' όλα ε, και ελπίζω ότι πράγματι θα προχωρήσουμε σε, μία, σε ένα κείμενο που να έχει σύνοχη να δίνει μια καθαρή εικόνα του πού θέλουμε να πάει η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να δώσει προβλεψιμότητα να είναι ρεαλιστικό και αρκετά ξεκάθαρο για την μεταβατική περίοδο μέχρι ότου επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει και ίσως θέσουμε και καινούργιους στόχους βάσει των νέων πηγών ενέργειας που μπορεί να βρίσκονται στην, ή να βρεθούν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Τζαβέλα. Ο κύριος Ρόιλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης εσά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω την εισηγήτρια, κάτι που κάνουμε τυπικά πάντοτε, αλλά στην περίπτωση αυτή το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση, διότι θεωρώ ότι η κυρία Τζαβέλα κατέβαλε τεράστια προσπάθεια σε πολλέ ε, πολλέ πολλές συνεργασίες, μια μεγάλη προσπάθεια για να συνοψίσει, να φέρει κοντά δηλαδή διάφορε απόψει που δεν είναι εύκολο διότι υπάρχουν πολλές πολιτικές ε, τοποθετήσεις πολύ διαφορετικές και ας το πω αυτό από την αρχή θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσέγγιση της συγκητρίας και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Αν όμως σε ορισμένα κεντρικά θέματα συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ίσως μπορούμε να θέσουμε σε ψηφοφορία δύο εναλλακτικέ συμβιβαστικές λύσεις, διότι δεν είμαι βέβαιος καν ότι με μια τροπολογία μπορούμε να καλύψουμε όλες τις απόψει της μια δικής μας πολιτικής ομάδας. Καμιά φορά τα θέματα αυτά της ενέργειας έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που διασπούν και τις ίδιε τι πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε αυτή την ελευθερία στου συναδέλφους. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να φτιάξουμε συμβαστικέ προτάσει, θαυμάσια. Αν όμω σε ορισμένα δεν είναι δυνατόν αυτό, τότε ίσως είναι σωστό να υπάρξουν και πλήρωνες τη μια συμβαστικές προτάσεις. Τώρα δεύτερο, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία ήταν, για παράδειγμα, το ερώτημα μπορούμε μακροπρόθεσμα να πούμε με ακρίβεια πώς θα εξελιχθεί κάποια προοπτική. Για παράδειγμα, αν εξετάσω την πολιτική της ενέργειας και του κλίματος των τελευταίων ετών, δεν είμαι και βέβαιος ότι πάντοτε ξεκινήσαμε από τις σωστές βάσεις ή ότι λάβαμε πάντα τις ε, σωστές αποφάσεις. Ορισμένες φορές λοιπόν είναι απαραίτητο να είμαστε και μετριοπαθείς και είναι σκόπιμο να φανούμε μετριοπαθείς και εμείς ως πολιτικοί και να μην θεωρούμε ότι με λίγες αποφάσεις που θα πάρουμε μέσα σε λίγα λεπτά θα σώσουμε τον κόσμο. Για παράδειγμα, η συζήτηση για δεσμευτικού στόχου και οι δεσμευτικοί στόχοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπω και η κυρία Τζαβέλα, είναι επιφυλακτικό απέναντι στην δεσμευτική στοχοθέτηση. Και δεν ξέρω πάλι αν είναι σωστό να επινοούμε διαρκώ νέου στόχου. Ίσως καλύτερα είναι να πούμε αν το σημαντικότερο είναι για, πολιτικά για μα να μειωθούν τα διοξίδια του άνθρακα, αυτό ας είναι ο βασικός μας στόχος θα δούμε μετά αν θα βάλουμε ίσως κάποιους υποστόχους ή ας πούμε μια έννοια όπως ορόσημα στην πορεία της επίτευξης των στόχων ή αν θα βάλουμε κάποιους επιμέρους στόχους για τις ανανεώσιμες ενέργειες, για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Αλλά να συνεχίσουμε απλώς να αυξάνουμε βάζοντας πάλι ένα 10% πάνω στους στόχους που κάποια στιγμή επινοήσαμε, βρίσκω ότι αυτό δεν είναι ούτε αποτελεσματικό ούτε ευφύες, διότι προφανώς δεν αποδίδει έχουμε και το πρόβλημα ότι με το εμπόριο, με την εμπορία μάλλον των εκπομπών, καμιά φορά στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε εκ παραλίλου τελικά οδηγούν στα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Πώς λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε μπορώ να επιτύχω αυτό που επιθυμώ με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ θα υποστηρίξω ευχαρίστως την κυρία Τζαβέλα. Βεβαίως μπορεί να προκύψουν εξελίξεις που αυτή τη στιγμή ίσως είναι αδιανόητες. Δέστε το σενάριο στην Αμερική. Με την απόφαση που έλαβαν για την εκμετάλλευση του shale gas ε, έχουν επαναστατικοποιήσει, αν μπορώ να πω έτσι, ολόκληρο τον κόσμο της ενέργειας στις ΗΠΑ. Με μια νέα πηγή ενέργειας που ξαφνικά ανεφάνει. Ανατροπή. Δεν χρειάζονται πλέον οι εισαγωγές ενέργειας απ' έξω. Καταφέρνουν και γίνονται ανεξάρτητοι. Πού ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει σε 20 ή σε 30 χρόνια, δηλαδή αν δεν θα προκύψει κάποια νέα πηγή ενέργεια ή κάποια νέα τεχνολογία. Έτσι λοιπόν έχω πολύ μεγάλη κατανόηση στην πρόταση να πούμε ρεαλιστική και αποτελεσματική. Πρέπει να είναι οι δρόμοι που θα ακολουθήσουμε. Η Κομισιόν πολύ καλά έκανε και μας αναγκάζει βάζοντας εναλλακτικά σενάρια ενώπιόν μας, μας αναγκάζει να σκεφτούμε με τον τρόπο αυτό με την έννοια ότι σήμερα με τη βάση που έχουμε τώρα αυτά μπορούμε να υπολογίσουμε. Αύριο μπορεί η βάση να έχει αλλάξει. Ο δικός χάρτης δεν είναι παρά η προετοιμασία για τη λήψη των αποφάσεων. Δεν είναι οι ίδιες οι αποφάσεις. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια βελτίωση ακόμη και συμπλήρωση με κάποια θέματα που ίσως λείπουν, αλλά στο τέλος θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια, όπως είπα, να μην θέλουμε, δε και καλά, με μία απόφαση να σώσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τα συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια. Έχουμε ήδη συναντηθεί και συζητήσει για, το, για τον φάκελο αυτό είναι σημαντικό θέμα διότι είναι προσανατολισμένο στο μέλλον. Και γι' αυτό χρειάζεται να το εξετάσουμε προσεκτικά. Ακόμη δεν μπορούμε να γνωρίζουμε βέβαια ποια μορφή θα έχει ο κόσμος το 2020. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το νέο τοπίο της ενέργειας, τι μορφή θα έχει λάβει. Αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα όραμα το 20-20-20 ή το 2030 διότι οι αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα θα έχουν βεβαίως απήχηση μέχρι το 2050. Είτε πρόκειται για τη δημιουργία υποδομών, είτε πρόκειται για τις, ε, για τις ε, ικανότητες, capacities δηλαδή. Αυτές οι αποφάσεις θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο 2050. Πρέπει να είναι σαφές βεβαίως ότι μέχρι τότε μπορεί να προκύψουν νέες τεχνολογίες πιο ε, ανεκτές από το περιβάλλον. Βεβαίως τότε θα τις χρησιμοποιήσουμε τις ε, τεχνολογίες αυτές. Οπωσδήποτε όμως το σύστημα ή τα συστήματα ενέργειας θα είναι πολύ διαφορετικά το 2050 και πρέπει να είναι εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για την προστασία του κλίματος. Αν θέλουμε επίσης να έχουμε μια ε, προμήθεια ενέργειας μέσα σε λογικό κόστος. Τι μας δείχνει η καθημερινή πράξη στην Ένωση. Μας δείχνει ότι όταν έχουμε δεσμευτικούς στόχους που μπορούν όμως να προσαρμόζονται με εύκαπτο τρόπο στις ανάγκες των χωρών μελών, όπως δηλαδή έχουμε στοχεύσει και στις ανανεώσιμες ενέργειες, τότε αυτές πραγματικά αποδίδουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν δεσμευτικούς στόχους που ωστόσο να μπορούν να ερμηνεύονται και με κάποιο εύκαμπτο τρόπο. Μου φαίνεται ότι δεν είναι λάθος να προβλέψουμε κάποιους ενδεικτικούς στόχους για το 2050. Στον οδικό της χάρτη η Κομισιόν έχει εξετάσει διάφορα σενάρια. Αυτό που βρίσκω σημαντικό και εντυπωσιακό μεταξύ των σενάριων αυτών είναι ότι ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για την πυρηνική ενέργεια ή ε, για την συμπαραγωγή. Ανεξαρτήτως λοιπόν των επιμερουστόχων στόχων, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια σχέση κόστους και τιμής. Δηλαδή πρέπει το κόστος να διατηρείται μέσα σε κάποια επίπεδα. Και εδώ πρέπει να γίνει μια σύγκριση, μια παραβολή των διαφόρων φορέων ενέργειας. και πρέπει να διασυνδεθούν οι προσπάθειες για την αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας με την προσπάθεια εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να αυξηθεί το ποσοστό των ανανεώσιμων ενεργειών με ε, ευρύτερο στόχο ίσως μέχρι το 2050 να βασιζόμαστε κυρίως σε αυτές. Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε ότι αυτό είναι το σενάριο που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσουμε. Η Κομισιόν νομίζω βέβαια έχει καλύτερη εποπτεία και αυτό είναι σημαντικό για τον οδικό χάρτη. Και επαναλαμβάνω ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι η δομή του κόστους. Εμείς νομίζω μπορούμε να πούμε τώρα στην Κομισιόν να κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς και να μπορέσουμε έτσι μετά να κάνουμε παραβολές μεταξύ των σενάριων. Εφόσον επιλέξουμε τις αναλώσιμες ενέργειες, θα πρέπει η Ένωση να παίζει ένα, ένα συντονιστικό ρόλο. Θα χρειαστούμε μεγάλα έργα, αλλά θα χρειαστούμε και πολλά μικρά έργα, τα οποία πρέπει να μπορούν να συνεπάρχουν στην αγορά. Και να μην λησμονούμε ότι ο κυριότερος, σημαντικότερος, ο κεντρικότερος παράγων είναι ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι πρέπει να πιστούν ότι από αυτούς εξαρτάται από την επιλογή των πηγών ενέργειας που θα κάνουν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χόλ. Η κυρία Χόλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, να την ευχαριστήσω θερμά διότι πραγματικά είχαμε με άκρο επικοδομητική συζήτηση και έγινε σκληρή δουλειά όχι μόνο από τους βουλευτές αλλά και από τους πολιτικούς συμβούλους για να καταλήξουμε σε συνένεση. Βέβαια δεν έχουμε ολοκληρώσει, ήδη Έχουμε όμως εντοπίσει τομείς ε, που πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε για το υψηλότερο επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Ένα σενάριο που λείπει και θα πρέπει πράγματι ε, αυτός ο κρίκος που λείπει να συνδεθεί, να προσθεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια σχετική ανάλυση. Όπως υπόθηκε, ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα είναι το κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το στόχο για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από το 2050 ή πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμη, γιατί ο στόχος διοξιδίου του άνθρακα σίγουρα ε, είναι απλός και αυτό τον καθιστά ελκυστικό στόχο, αλλά υπάρχουν προβλήματα, διότι το να μιλάμε μόνο για διοξίδιο του άνθρακα. Πρόκειται για έναν αρκετά χαλαρό και θα έλεγα κάπως αναξιόπιστο στόχο. Συζητήσαμε και το ETS ε, για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών και ξέρουμε ότι η τιμή του άνθρακα δεν δίνει τα μηνύματα που πρέπει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες όπως η κρίση για παράδειγμα που έχουν επηρεάσει αυτό το σύστημα και κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση την τιμή του άνθρακα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τους στόχους μας για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όχι μόνο γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την οικονομική κρίση, αλλά και γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να εκπληρώσουμε τους στόχους μας για το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά με βελτιωμένη οικονομία και με προοπτικές ε, ευημερίας, ανάκαμψης. Ε, ας είμαστε αισιόδοξοι, να μην θεωρούμε ότι το 2030, πόσο μάλλον το 2050 θα είμαστε ακόμα σε κρίση οικονομική. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα θα δώσει τόσα κίνητρα στην ε, βιομηχανία για να επενδύσει. Νομίζω ότι πρέπει όλους τους στόχους να τους λάβουμε υπόψη, όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Η ο κλάδος των ανανοσίμων νομίζω ότι έχει γνωρίσει πρωτόγνωρη ανάπτυξη, άνοδος της τάξης του 6% ετησίως παρατηρείται στον τομέα αυτό. Είναι πάρα πολύ καλή απόδοση ε, του κλάδου αυτού. Δημιουργεί θέσει εργασία. Ακόμη και σήμερα που έχουμε κρίση, οι ε, άνθρωποι, οι επιχειρήσει που επενδύουν όμω, θα πρέπει να ξέρουν πού βρισκόμαστε μετά το 2020. Διότι αλλιώ αυτό το νέο τομέα ανάπτυξη κινδυνεύουμε να τον δούμε να ε, τελματώνει ή να σημειώνει ύφεση αφού δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά το 2020. Ακούω ε, και ξέρω ότι στο γεύμα συζητήθηκε και η βιομηχανική πολιτική από το Επιτρόπο Ταγιάννη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε έναν τομέα βιομηχανικής πολιτικής που τα πηγαίνει περίφημα αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να δίνουμε ε, τα σωστά σημάδια στους επενδυτές. Και ένας άλλος τομέας που πρέπει να συμπεριληφθεί είναι η ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία μας. Δεν τα πήγαμε καλά με τους στόχους του 2020. Λένε πολλοί ότι α, τα κράτη-μέλη ούτω ή άλλω θα ασχοληθούν με την ενεργειακή απόδοση και δεν το έκαναν ή το ξέχασαν γιατί δεν ήταν όλα αυτά πολύ ξεκάθαρα ορισμένα. Ιδίω στον τομέα των οικοδομών υπάρχουν οδικοί χάρτε για τη φυστάμενα κτίρια, αλλά πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομική αποδοτικότητα. Και να μην δαπανάμε τόσο πολύ ενέργεια, είτε είναι ανάσχημες είτε άλλη. Τέλος, για το αέριο. Έχουμε πάρα πολλές ε, φιλοδοκ... μάλλον έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ε, προσδοκίες ε, το ενδεχόμενο ε, εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού αερίου. Αλλά ε, θα μπορέσουμε να απεμπλακούμε πλήρως από τον άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρισμού μέχρι το 2030. Και αν διαβάσει κανείς και τι λέει και η Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή και δεν χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας πολιτικά επιχειρήματα. Θα πρέπει σίγουρα να βρεθεί μια επανεξισορρόπηση του όλου συστήματος παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2030. Αν το φυσικό αέριο θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργειακού μείγματος, αυτό θα πρέπει να συνδεστεί και με την ε, συγκράτηση του, και αποθήκευση του άθρακα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ε, πώς θα είναι τα πράγματα. Ίσως χρειαστεί να παραμείνει μέσα στο υπέδαφος το, το αέριο. Και κάτι ακόμη, σε ό,τι αφορά τις τιμές, Δύο πράγματα που συχνά ξεχνούμε είναι πρώτον ότι η αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων ουσιαστικά συμβάλλει στην αύξηση των τιμών κατανάλωσης. Και δεύτερον, η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας πρόσφατα είπε ότι 66 δις επιδοτήσεων πήραν το 2010 οι ανανεώσιμες ε, πηγές, ενώ τα ορυκτά 409, έξι φορές παραπάνω δηλαδή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Presidenta. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια κυρία Τζαβέλα για τη δουλειά της αλλά και για τη στάση της, διότι πάντοτε ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη, ε, ανοιχτή προς απόψη όλων των ε, βουλευτών, συναδέλφων. Η έκθεση αυτή δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι μας δίνει την δυνατότητα να σκεφτούμε την ενεργειακή μας στρατηγική για το μέλλον, μετά δηλαδή από το 2020. Η ενέργεια απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, άρα και μακρόπνοη στρατηγική και η ενεργειακή πολιτική επίσης είναι τέτοιας φύσης, τέτοιας φύσης που πολλές φορές ε, καθυστερεί, περνάει χρόνος να καταλάβουμε τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά που να τα υπόψη μας, γι' αυτό πρέπει να έχουμε και έναν πιο μακρό χρονικό ορίζοντα στο μυαλό μας. Αυτή η στρατηγική, συμφωνούμε όλοι, ότι θα πρέπει να έχει ως στόχο την ασφάλεια του εφοδιασμού, που θα πρέπει να είναι και ανταγωνιστικός ε, και βιώσιμος και πάντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλες τις πηγές, όλες τις τεχνολογίες και αυτέ που έχουμε ήδη στη θέση μας και άλλε που θα μπορούσαν να προκύψουν και θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Πολλοί συνάδελφοι όμως πιστεύουν ότι αυτή η σκέψη πρέπει να είναι ουδέτερη κατά κάποιο τρόπο και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ιδέα ε, για έναν νέο στόχο μείωση των εκπομπών. Αυτός ο ε, νέος στόχος, ο μόνος στόχος αν θέλετε, πρέπει να είναι κίνητρο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργεια αλλά και για μέτρων ενεργειακή απόδοση. Χωρί όμω να αποκλεί άλλε πηγέ, όπω σχιστολιθικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, που αντιπροσωπεύουν και αυτές ε, ένα θετικό ε, στοιχείο σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι υπάρχει και εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε, αλλά δεν το καταφέρνουμε. Πόρα απέχουμε μάλιστα. Και πρέπει να στρέψουμε και το βλέμμα μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι οι Ευρωπαίοι πολλές φορές είμαστε λίγο και ευρωκεντρικοί. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε και τις άλλες ε, περιοχές του κόσμου. Όταν σε άλλες χώρες αναδύεται μια νέα τεχνολογία, ιδίως όταν με τις ενέργειες, εκεί βλέπουν τι δυνατότητες ε, διανοίγονται, ενώ εμείς βλέπουμε μόνο κινδύνους και προβλήματα. Αλλά κάθε τεχνολογία έχει κινδύνους, αλλά έχει και πλεονεκτήματα, έχει και ευκαιρίες, δυνατότητες. Ενώ εμείς επικεντρωνόμαστε μόνο στα προβλήματα, στους κινδύνους, στις δυσκολίες και αυτό μας παραλύει. Άλλες χώρες εστιάζουν πολύ περισσότερο ε, και με μεγαλύτερη τόλμη θα έλεγα στις ευκαιρίες και όχι στον κίνδυνο. Αν δούμε και τι έγινε στη διάσκεψη της ε, Ντόχα, πράγματι υπήρξαν σημαντικές ε, απογοητεύσεις ε, με κάποιες χώρες όπως είναι η Ιαπωνία, ο Καναδάς. Είδαμε τι έκαναν επίσης η Κίνα, η ΙΠΑ ή τι δεν έκαναν. Ε, εμείς ε, πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε ένας μέτριος, μετροπαθής παράγοντας στον τομέα των εκπομπών. Η συμβολή μας μπορεί να είναι υποδειγματική, μπορεί να είναι αξιέπαινη. Αν είμαστε μόνοι μας, δεν θα είναι και τόσο χρήσιμη. Επομένως, ενοιολογικά μας έχει βοηθήσει η κυρία Τζαβέλα να θεσπίσουμε αυτό το πλαίσιο, αλλά πρέπει να δούμε τελικά αν θα πετύχουμε να έχουμε μια έκθεση όπου όλα αυτά τα ζητήματα θα περιλαμβάνονται και αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θέση για αυτή την μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν θα είναι ομόφωνη, είμαι ε, βέβαιο, αλλά, πιστεύω θα τη στηρίξει η ευρύτατη πλειοψηφία. Αυτό τουλάχιστον είναι ο στόχο μας. Σας ευχαριστούμε κυρία Κολάσκα Πουμπίνσκα. E, e, Ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερος για την εργασία της κυρίας Τζαβέλα. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση είναι πάρα πολύ καλή. Και διότι, βεβαίω το λέω αυτό και διότι είμαι εισηγήτρια, αλλά διότι περιλαμβάνει ορισμένες ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Και ιδίω εφόσον ε, μιλούμε για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να μιλήσουμε και για τους μεταστόχους, που σημαίνει ότι μιλούμε για την περαιτέρω οικονομική εξέλιξη της Ευρώπης, μια ισορροπημένη εξέλιξη η οποία πρέπει να βασίζεται και σωστή ενεργειακή ε, λύση. η αλλαγή του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης, αλλά και των κλιματικών στόχων, αλλά επίσης ένα σημαντικό ρόλο παίζει και η ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. Είναι όλοι αυτοί οι στόχοι τους οποίους πρέπει να συζητήσουμε και είναι οι στόχοι που πρέπει να είναι ισορροπημένοι μεταξύ τους τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα απαιτήσει κάποια ευκαμψία εκ μέρους μας και ένα πνεύμα ανοιχτό. Και γι' αυτό συγχαίρω για την ε, έκθεση. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η στρατηγική αργότερα θα ε, εφαρμοστεί στις περιφέρειες από διάφορους φορείς. Είναι πολύ διαφορετικές οι οργανώσεις, οι οργανισμοί, οι αρχές αυτές έχουν και πολύ διαφορετική γεωγραφική κατανομή. Αν λοιπόν φτιάξουμε ένα ενιαίο πρότυπο για όλη την Ευρώπη, πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη όλη αυτή την ποικιλία ιδιαιτεροτήτων. Γι' αυτό και επιθυμώ στην έκθεση να περιληφθούν και οι συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας που προσέφερε υπηρεσίες στην Επιτροπή Σχεδιασμού και η οποία είπε ότι σε κάθε σενάριο πρέπει να περιλαμβάνεται ένα στοιχείο συνέργειας έτσι ώστε να τονιστεί και η ανάγκη περιορισμού των εκπομπών οξυδίων του άνθρακα και ότι όλοι οι στόχοι εξυπηρετούνται από τις προσπάθειες όλων των περιφερειών. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται προσαρμογή των στόχων. Σας ευχαριστώ κύριο Σάρις Βόλσκα. Molto grazie, Presidente. Ah, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνο ε, για την ε, τοποθέτηση τη Επιτροπή ΑΘΕΤ ε, σε σχέση με την έκθεση τη κυρία Νταπέλα. Να την ευχαριστήσω λοιπόν για την διεξοδική έκθεση και που έλαβε υπόψη της την θέση της ΑΘΕΤ, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα σχεδόν από τα μέλη της Επιτροπής ΑΘΕΤ. Τώρα η ουσία της δικής μας τοποθέτησης. Κατά πρώτον, θεωρούμε ότι η ενεργειακή πολιτική είναι μια αυτόνομη πολιτική με εξίσου σημαντικέ διαστάσεις όπως ε, η εξωτερική πολιτική. Όμως είναι μια αυτόνομη πολιτική και όχι ένα παραπροϊόν της πολιτικής μας για τις κλιματικές αλλαγές. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θέλουμε να δοθεί έμφαση στις γεωπολιτικές επιπτώσεις και το διεθνές, το, το αντίκτυπο στις διεθνείς μας σχέσεις που έχει η στρατηγική για το 2050. Γι' αυτό κάναμε κάποια αποκριτικά σχόλια για κάποιες προτάσεις, καθώς το έγγραφο δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη την πολιτική διάσταση της ενεργειακής στρατηγικής. Όπως είπα, υπάρχει εξωτερική αυτή συνιστόσα. Δεν είναι απλώς ένα προϊόν η ενέργεια, είναι ένα πολιτικό εργαλείο στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αν όχι ένα όπλο. Ο, δικός, ο χάρτης πορείας, ειδωμένος από αυτή τη σκοπιά, χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις. Είναι υπεραισιόδοξο να πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για τι κλιματικέ αλλαγέ βάσει των όρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι το θετικότερο σενάριο ότι οι υπόλοιποι εταίροι μα παγκοσμίω θα δεχτούν του δικού μα όρου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια δεύτερη επιλογή, ένα plan B όπως λέμε, για να διασφαλίσουμε την ενεργική μας ανεξαρτησία και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι νέε ευκαιρίες και οι δρόμοι για την αναφοδιασμό μας, όπως το σχιστολιθικό αέριο, ένα νεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να έχουμε μια σφαιρική θεώρηση και ω προ τη διάσταση τη εξωτερική πολιτική και τη ε, πολιτική των εμπορικών μα σχέσεων. Δεν πρέπει να βλέπουμε την ενεργειακή πολιτική ω παραπροϊόν τη πολιτική για τι κλιματικέ αλλαγέ. Στο άμεσο μέλλον θα παραμείνει ένα εργαλείο τη εξωτερική πολιτική η ενεργειακή πολιτική. Θα δεχτούμε πιέσει από του εταίρου μα και ό,τι και να γίνει πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα ενεργειακή ασφάλεια που να συμπεριλαμβάνεται σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε και τι συμφωνίε εταιρική συνεργασία ή σύνδεση με τρίτε χώρε θα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας ε, συμπεριφοράς και να, ε, δίδεται, να δίδεται έμφαση στα μέτρα ε, που θα λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπίζονται μονομερείς μεταβολές τάσεις από τους εμπορικούς μας εταίρους. Είναι κάπως θετική η προσέγγιση της έκθεσης, διότι δεν λαμβάνει υπόψη τους αναδυόμενους παραγωγούς, τις νέες τεχνολογίες, τις νέες ροές ζήτηση και προσφοράς, ακόμη και τις ασύμβατες πηγές άντλησης ενέργειας, οι ε, Αρκτική και η Μεσόγειος. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος να παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους. Η τοποθέτηση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, δίνει έμφαση στο ότι η Ευρωπαϊκή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να εξάγει το ρυθμιστικό πλαίσιο τη και σε τρίτες χώρες και χρησιμοποιώντα τα εργαλεία που ήδη διαθέτει. Όπω το τρίτο ενεργειακό πακέτο για την ενέργεια, την σχετική συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια και για την ενέργεια γενικότερα. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν μαζί μας οι εταίροι μας ε, για να μην αντιμετωπίζουμε απρόβλεπτες απειλές όπως συμβαίνει τώρα με τη Μολδαβία και τη Ρωσία και την Κάσπρομ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ενισχύσει εδώ την Μολδαβία, δίδοντα όχι μόνο δυνατότητε μετάβαση ή εξαιρέσει, όπω έχει κάνει με τη Μολδαβία για το τρίτο ενεργειακό πακέτο, αλλά και με μια συνολική δεσμή μέτρων, όπως το να κάνει συστάσεις προς τους εταίρους της Μολδαβίας, να υιοθετήσουν το δικό μας κεκτημένο και να ε, έχουν διασυνδέσεις με άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ρουμανία δηλαδή, που είναι πολύ κοντά χιλιομετρικά στην ε, Μολδαβία. Η ανεξαρτησία μας ενεργειακά μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διεύρυνση της ενεργειακής μας πολιτικής στα ανατολικά και νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως και ένας άλλος στρατηγικός στόχος που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ποικιλομορφία της ε, παροχής και των δρόμων τη ενέργεια και αυξάνοντας την ασφάλεια του νότιου ε, διαδρόμου λόγου χάρη, Southern Corridor, που δεν πρέπει όμως να τον ε, συγχαίουμε με τον ε, νότιο αγωγό, διότι δεν θέλουμε να υπάρξουν εξαιρεσει όπως αυτές του Nord Stream ε, για τη Ρωσία πρόσφατα. Για το Αζερβαϊτζάν και άλλες ε, χώρες εταίρους μας υπάρχει ανυπομονησία. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εντολή να διεξαγάγει διαπραγματεύσει για τη στατηγική ε, διαφοροποίηση των προγραμμάτων τη Ένωση προ την ενέργεια για τον αγωγό που θα διασχεί την Κασπία και τις συζητήσεις με το Τουρκμενιστάν και το Αζερβαϊτζάν χρειάζονται εντατικοποιημένες συνομιλίες, διαφάνεια, συντονισμός και αποτελεσματικότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται να γίνουν, να γίνουν βήματα προόδου ώστε να έχουμε καλύτερη προμήθεια εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γνωμοδότηση δίνει έμφαση και στι σχέσει μα για την ενέργεια με τη Ρωσία, ε, καλώντα να δημιουργηθεί ένα οδικό χάρτη ε, για τι σχέσει αυτέ ε, για το μέλλον και να δοθεί έμφαση στην αμοιβαιότητα καθώ και τη συμφωνία για την ενέργεια, τη χάρτα για την ενέργεια και το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Χρειάζεται μια ε, συνεκτική υλοποίηση των ε, σχετικών όρων και του δικαίου για την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα σε όλε αυτέ τι χώρε που λειτουργούν βεβαίω εκτό ε, τη επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω η Gazprom, αλλά επικουρικά καλύπτουν τι δικέ μα ανάγκε. Επίση, καλούμε όλε τι εταιρείε που λειτουργούν στον τομέα τη ενέργεια να συνεργαστούν με τις ερευνητικές αρχές, άσχετα με αυτό που ζητήθηκε από το διάταγμα του Πούτιν, και να αναλυθεί δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σχετικά προβλήματα. Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους όλους τους σκιώδεις εισηγητές από την Επιτροπή μου και τον κύριο Ρόιλ και την κυρία Ζαβέ, Τζαβέλα βεβαίως την ίδια για την ε, πολύ συνολική της προσέγγιση. Σας ευχαριστούμε. Grazie. Ευχαριστούμε. Αφήσαμε λίγο περισσότερο χρόνο στον συνάδελφο Σάριο Βόλσκι γιατί μας παρουσίασε τη θέση τη δική του επιτροπή. Ε, τώρα το κ. Κρότσμαν. Κ. Κρότσμαν, ευχαριστώ. Επιθυμώ να τονίσω μία πτυχή που δεν περιλαμβάνεται στον οδικό χάρτη και εννοώ την δημογραφική εξέλιξη. Εάν στη Γερμανία έχουμε 20 εκατομμύρια λιγότερους, θα έχουμε και 20 εκατομμύρια λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερη ανάγκη χρήσης ενέργειας για τα σπίτια και δεν ξέρω και ποια είναι τα νούμερα για ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει δίκιο κατά τούτο ο κύριος Ρόιλ ότι χρειάζεται προσαρμογή στη χρονική εξέλιξη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει σε 10, 20, 30, 50 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε σε κάποιους στόχους, είτε πρόκειται για μείωση των οξυδίων του άνθρακα ή για τις ανανόσιμες ενέργειες, αλλά οι στόχοι αυτοί να είναι ρεαλιστικοί και προσαρμόσιμοι. Επίσης εδώ τονίζω ότι σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη και η δημογραφική εξέλιξη, η οποία θα οδηγήσει στο ότι θα χρειαζόμαστε λιγότερη ενέργεια. Και γι' αυτό οι στόχοι μας πρέπει να εκτιμηθούν με ρεαλισμό και να είναι υλοποιήσιμοι και να μην βλάψουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Διότι ακόμα υπάρχει πολλής δρόμος μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το 20% του ΑΕΠ που λέει ο ε, Επίτροπος. Ευχαριστούμε κύριε Κρόιτσμαν. η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you. Ευχαριστώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μας προς την κυρία Τζαβέλα και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για αυτό το σχέδιο έκθεσης που καλωσορίζουμε. Είναι μια ουσιαστική συνεισφορά στην όλη συζήτηση που θέλαμε να διοργανωθεί στα πλαίσια του χάρτη πορείας για το 2050 για την ενέργεια. Να σταθώ σε μερικά σημεία που μας απασχολούν. Πρώτα απ' όλα είναι αλήθεια ότι ε, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιε προβλέψει βάσει όμω συγκεκριμένων δεδομένων. Γι' αυτό καταρτήσαμε κάποια σενάρια και να δούμε ποιο ήταν ο αντίκτυπο αν κάνουμε τη μια ή την άλλη επιλογή. Ποιο ήταν ο αντίκτυπο στι τιμέ, στην εξάρτησή μα από τι εισαγωγέ και σε άλλα ζητήματα. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια δεν επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον σενάριο, συνδυάζοντα τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όμω, όπω είπα προηγουμένω, η υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, το σενάριο δηλαδή αυτό, ε, περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών. Πάντω και οι πέντε, τα πέντε σενάρια που δημιουργήσαμε ε, λαμβάνουν υπόψη τη μείωση ενέργεια ε, ω το 2050 με ένα ελάχιστο ποσοστό του 38%. Αυτό είναι βασικός πολιτικός στόχος. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την ενεργειακή αποδοτικότητα αν θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας. Επίσης, να συμφωνήσω ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις προσπάθειές μας. Το είπε ο κ. Ρόιλ και άλλοι ε, βουλευτές. Ο κόσμος, το σκηνικό της ενέργειας ε, μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς. Ε, υπάρχουν και άλλα σενάρια αναφοράς βασικέ αρχέ δηλαδή για το μελλοντικό μα έργο που ανανεώνεται τριετία. Χρησιμοποίησαμε εδώ τα δεδομένα που είχαμε από το 2009, αλλά βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία των συζητήσεων με τα κράτη-μέλη για τον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των κλιματικών αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και τις μακροοικονομικές, γεωγραφικές, γεωπολιτικές εξελίξεις και το νέο σενάριο αναφοράς που δημιουργούμε, ε, λαμβάνοντας υπόψη και το αέριο, το σέλγκας, ε, που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό μας σενάριο πριν από δύο χρόνια, γιατί αυτό δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, τώρα το περιλαμβάνει λοιπόν το σενάριο αυτό αναφοράς, το οποίο θα δημοσιευτεί την Άνοιξη. Εκεί θα αντικατοπτρίζονται όλες οι πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο. Και τέλο, θα το έθιξε αυτό η κυρία Τζαβέλα, η συζήτηση για τον ε, χάρτη πορεία για το 2050 είναι βάση των εργασιών μα για την ερχόμενη χρονιά. Έχουμε ένα πρόγραμμα εργασία με μια δεσμή μέτρων για την ενέργεια και τι κλιματικέ αλλαγέ για το 2030 και βεβαίω χρειαζόμαστε περισσότερε προβλέψει, περισσότερη σαφήνεια και θα μελετήσουμε τα διάφορα σενάρια, το έργο που ήδη έχει γίνει και τις όλες τις συζητήσεις, το διάλογο που είχαμε ως βάση για ε, την ερχόμενη φάση και το πολιτικό πλαίσιο την Άνοιξη για το 2030 θα περιλαμβάνει ένα σχετικό έγγραφο βάση διαβουλεύσεων όπου θα πρέπει να προχωρήσουμε γρηγορότερα, να δούμε αν θέλουμε δεσμευτικού στόχου, εάν θα παραμείνουμε στο στόχο του 2020, αν θα του αλλάξουμε και θα περάσουμε σε κάτι καινούριο. Είναι ανοιχτή ακόμη η συζήτηση, γι' αυτό η συνεισφορά σα είναι πολύτιμη. Θα φροντίσουμε η συζήτηση αυτή να συνεχιστεί και του χρόνου, περιλαμβάνοντα και μια αξιολόγηση για το πώ έχουμε πάει ω τώρα σε σχέση με του στόχου του 2020. Πώ συσχετίζονται οι στόχοι αυτοί με του επόμενου και ελπίζουμε ότι του χρόνου από την πλευρά της Επιτροπής θα έχουμε ετοιμάσει κάτι που μπορούμε, να μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε με τον ορίζοντα του 2030. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε. Και τώρα κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος και ευχαριστώ όλους με την συνεισφορά του στη σημερινή συζήτηση. Ε, από ό,τι βλέπω επικεντρωνόμαστε στο θέμα των στόχων και συμφωνώ ότι πρέπει να είναι ρεαλιστική, υλοποιήσιμη και προσαρμόσιμη. Ε, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για να δείτε ότι πράγματι ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ε, αισιόδοξε προβλέψεις. βλέπω ότι οι οπαδοί των ανανεώσιμων πηγών έχουν μια πολύ θετική άποψη. Σας ενημερώνω ότι στη χώρα μου, η οποία ενδείκνυται για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από, από τον τοπικό πληθυσμό στην εγκατάσταση των, ε, ανεμο, των φωτοβολταϊκών πρώτα απ' όλα ε, αλλά επίσης και τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή όταν είναι μια χώρα η οποία έχει μικρά νησιά με τουρισμό και τα λοιπά και πάμε και, κα... Ε, και τοποθετούμε νεμογεννήτριες υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίδραση. Αντίδραση λοιπόν στις ανανεώσιμες υπάρχει και δεν θα πρέπει να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι οι ανανεώσιμες πηγές θα μας βοηθήσουν να πιάσουμε τους στόχους. Να έχουμε στόχους υλοποιήσιμους, ρεαλιστικούς να περιγράψουμε τη μεταβατική περίοδο και υιοθετώ και αυτό που είπε ο κύριος Κουάνδρας, να είμαστε θαραλέοι ως Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη έχει δικά της αποθέματα, δικό της πλούτο και δεν μπορούμε να στερούμε τους λαούς της Ευρώπης από την αξιοποίηση του πλούτου της. Με το να λέμε ότι να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε ενεργειακή πηγή πλην των ανανεώσιμων ως απειλή νομίζω ότι είναι θα έλεγα μια βαριά κουβέντα είναι ντροπή για την Ευρώπη είναι πρόκληση δεν είναι απειλή ό,τι το θεωρούμε ότι είναι ίσως επικίνδυνο να επιδιώξουμε να το κάνουμε ακίνδυνο η Ευρώπη πρωτοπόρησε σε όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει πίσω και να λέει ότι όχι, το θεωρώ αυτό ως απειλή για την κλιματική αλλαγή, δεν το υιοθετώ. Είναι πρόκληση και θα πρέπει με την τεχνική υποστήριξη και με τις νέες τεχνολογίες πράγματι να βρίσκουμε τους τρόπους να αξιοποιήσουμε τα ενεργειακά μας αποθέματα. Ελπίζω και προσδοκώ σε πράγματι μια καλή ε, συνεργασία. Το θέμα των στόχων θα τον περιγράψουμε μέσα σε αυτά τα οποία υπόθηκαν από όλους σας και νομίζω ότι θα βρούμε μια ε, λύση αλλά θα ήθελα όλοι να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα κείμενο το οποίο να έχει συνοχή και να ανταποκρίνεται σε μια Ευρώπη 27 κρατών, όχι τριών ή πέντε ή οκτώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Γρία Τζαβέλα. Κλείνουμε τη συζήτηση αυτή. Θυμίζω ότι η προφορία στην Ήτρε θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια το θέμα θα περάσει τον Μάρτιο του 2013. Τώρα να περάσουμε στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Ούλφ όμως θα ξεκινήσουμε την ε, σχετική συζήτηση με μία παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που για 15 λεπτά θα μας παρουσιάσει τη δική της ε, οπτική για το θέμα. Um, thank you very much, uh, Chair. Um, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τον κανονισμό για την ηλεκτρονική αναγνώριση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσω να μείνω στο 15 λεπτό που όρισε η Πρόεδρος όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Κομισιόν ενέκρινε ε, μια ανακοίνωση για την ηλεκτρονική αναγνώριση και υπηρεσίες εμπιστοσύνη για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στις 4 Ιουνίου του 2012. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια πρόταση που αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην υλοποίηση τη ψηφιακή ατζέντα, ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και το δικό χάρτη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Που πολύ ε, σωστά θεώρησε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μία από τι βασικέ 12 fast track ε, δράσει. Στόχο είναι να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό τη ε, διαδικτυακή επανάσταση. Θέλουμε επίση να παράσχουμε ένα αξιόπιστο ασφαλέ περιβάλλον που θα ανοίξει την πόρτα σε διασυνοριακές ασφαλείς όμως υπηρεσίες και θα δημιουργήσει επίσης και θέσεις εργασίας, ανάπτυξη για να ανθίσει η ενιαία αγορά στην Ευρώπη. Η πρόταση λοιπόν έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενίας αγοράς, τονώνοντας την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στις διασυνοριακές. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Η πρότασή μας λοιπόν έχει ως στόχο και οι ιδιώτες αλλά και οι επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, τις ε, εθνικές ηλεκτρονικές του ταυτότητες και διασυνοριακά για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες, τουλάχιστον δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Συμποθέσουμε υποθέσουμε ότι μια φοιτήτρια από το Βέλγιο, η Ελίσσα, θέλει να γραφτεί σε ένα Ιταλικό πανεπιστήμιο θα μπορεί να κάνει όλες τις σχετικές διαδικασίες online, χρησιμοποιώντας για αναγνώριση τη βελική της ταυτότητα, ηλεκτρονική ταυτότητα. Και θέλω να καταστήσω πως ότι αυτό δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Έχουμε ήδη κάνει μια πιλωτική, ε, μάλλον σειρά πιλωτικών προγραμμάτων και πρόσφατα και αποδείξαμε ότι μπορούν αυτά τα συστήματα να λειτουργήσουν. Είναι καινοτόμοι τρόποι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης και να, είναι πολύ, να διευκολύνουμε τις ε, δημόσιες συναλλαγές μας. Πριν αναφερθώ πιο πολύ στο περιεχόμενο, θέλω να πω τι δεν θα καλύπτει ο κανονισμός. Δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ηλεκτρονική ταυτότητα ή άλλα προγράμματα ηλεκτρονικής ε, ταυτοποίησης ή αναγνώρισης. Απλά αποσκοπεί η πρόταση αυτή σε αυτές τις χώρες που υπάρχει ηλεκτρονική αναγνώριση να μπορεί να χρησιμοποιείται διασυνοριακά αλλά με πλήρη σεβασμό στου κανόνε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίση, δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη αυτή η πρόταση να κοινοποιούν τα προγράμματα που έχουν για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση να μην τα κοινοποιούν στην Κομισιόν υποχρεωτικά. Ούτε προτείνει τη δημιουργία μιας καινούρια ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής ταυτότητας ή κάποιας βάσης δεδομένων ε, ευρωπαϊκής. Πώς θα λειτουργεί λοιπόν. Ουσιαστικά θα έρει αυτή η πρόταση τα προβλήματα και έτσι θα μπορεί να παρέχει συνεχείς και αδιάλειπτες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που θα έχουν την ίδια νομική αξία όπως και παραδοσιακές ε, διαδικασίες ή έντυπες. Το ίδιο λοιπόν θα γίνεται και με τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Έχουμε και τις ηλεκτρονικές φραγίδες, έχουμε χρονοσφραγίδες ε, και άλλα ε, αποδοχή ηλεκτρονικών εγγράφων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούν να γίνουν και θα αναγνωρίζονται και θα υπάρχει ένα ε, πρότυπο για την ασφάλεια δικαίου. Θα μπορούμε έτσι να εμπιστευόμαστε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και έτσι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα οι χρήστες, θα είναι πιο εύκολη η πρόσβασή τους και θα είναι και μεγαλύτερη και εμπιστοσύνη σε αυτές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα νομικά ασφαλές περιβάλλον και αξιόπιστο για τη χρήση αυτών των ε, υπηρεσιών. Και με αυτή την πρόταση θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έδειξε η ανεπιτυχής εφαρμογή της οδηγίας ηλεκτρονικής ε, υπογραφής του 99 που δεν δημιούργησε τελικά ένα αρμονισμένο νομικό και τεχνικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ούτε τόνωσε την ανάπτυξη δεσυνοριακών αγορών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα για να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Υποθέσουμε ότι έχουμε μια γαλλική εταιρεία, εταιρεία σε μέτρα τη Γαλλία που θέλει να, που παρέχει συμβάσεις. Έχουμε έναν ομόλογο στη Γαλλία και έναν άλλο σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτά θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά όλες οι συναλλαγές Με την πρόταση αυτή λοιπόν δίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για όσου χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση και ηλεκτρονικέ υπηρεσίε εμπιστοσύνη όπω ηλεκτρονική υπογραφή. Επίση, θα παρέχει καλύτερε επιγραμμικές σε υπηρεσίε. υπηρεσίες γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Θα είναι πιο βολικέ οι δημόσιε υπηρεσίες και βέβαια η πρόταση αυτή θα εξοικονομεί και χρόνο και χρήμα για του πολίτε και τι επιχειρήσει. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα βελτιώσει και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Παραδείγματο χάρη για πρόσβαση στι κρατικέ υπηρεσίε ή σε διαγωνισμού σε άλλων χωρών. Τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό θα είναι ότι θα μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού, άρα φιλοπεριβαλλοντικό το μέτρο. Θα έχουμε λοιπόν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε που θα είναι και πιο εύκολε και έτσι οι χρήστε θα έχουν την ασφάλεια δικαίου που θα τους κάνει να επιλέγουν ε, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις ολοκληρώνουν με ασφάλεια και με εύκολο τρόπο. Εν συντομία τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω και για τις οικονομικές επιπτώσεις ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ε, έχουμε διάφορες μελέτες, εγώ θα αναφερθώ μόνο στην ανάλυση Μάικος Κονσάλτ που λέει ότι για την ολοκλήρωση ψηφιακού περιβάλλοντος θα έχουμε 4% ανάπτυξη του ποσοστού επί του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν σημαντικά ωφέλη, άρα πρέπει να ολοκληρωθεί η νέα ψηφιακή αγορά. Είναι σημαντικός στόχος. Και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε δεν θα πρέπει να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποιες διατάξεις της ηλεκτρονικής υπογραφές. Έτσι, ο προτινόμενος κανονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την καλή λειτουργία σημαντικής κλαδικής νομοθεσίας όπως οδηγία για τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, ηλεκτρονική τιμολόγηση, πρωτοβουλία πολιτών, επειδή όλα αυτά βασίζονται στις ηλεκτρονικές υπογραφές. Ποιος θα ωφεληθεί λοιπόν από την πρόταση αυτή, όπως σας είπα, είναι σαφές μεν και μπορεί κανείς να το καταλάβει ότι οι πολίτες είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν. 100.000 περίπου φοιτητέ οι οποίοι μετακινούνται, ε, πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Πρέπει να ε, αλλάξουν τη διεύθυνσή τους, να ε, επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Θα μπορούν πάρα πολύ εύκολα να το κάνουν ηλεκτρονικά επιχειρήσει θα ωφεληθούν επίσης και αυτό αυτονόητο. Η πρόταση είναι πολύ σημαντική γιατί θα δώσει τη δυνατότητα διασυνοριακής επιχειρηματική δράσης. Πιο, ε, μεγαλύτερη διευκόλυνση των διοικητικών υπηρεσιών. Λιγότερο χαρτομάνι, περισσότερη επιτελεσματικότητα, λιγότερο κόστος. Ένα παράδειγμα. Έχουμε μία πύλη στην Εστονία, Registration Portal, μέσω της οποίας αυτής πύλης μπορεί μέσα σε 8 λεπτά μια εταιρεία μπορεί είτε με την χρήση της εστονικής ταυτότητας ή στο μέλλον με χρήση βελγικής, πορτογαλικής, λιθουανικής να να μπορέσει να ιδρύσει μια εταιρεία περιορισμένη ευθύνη. Και θα μπορεί επίση ε, ο ισολογισμό μια εταιρεία ε, επίση πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 20 λεπτά ηλεκτρονικά να μπορεί να καταρτιστεί. Πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, δυνητικές. Ένα σημαντικό παράδειγμα θα ήθελα να σας δώσω για το πόσο μπορεί να επηρεάσει οικονομικά αυτός ο κανονισμός. Στον τομέα των ηλεκτρονικών τιμολογίων, από το να περάσουμε στο χαρτί στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, θα έχει αποτέλεσμα από 8,6 ευρώ ανά τιμολόγιο να πέσει το κόστο στα 2 ευρώ περίπου. Μείωση του κόστου κατά 80% περίπου δηλαδή. Γιατί λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά κάνει τη διαφορά αυτός ο κανονισμός. Γιατί προσφέρει μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία μέσων ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνη, Επίσης, ενισχύει τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίηση, που βοηθά και διευκολύνει τι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ένα σημαντικό ε, κομμάτι για τη δημιουργία της ε, ενιαίας αγοράς για την πολύ σημαντική οικονομική αυτή περιοχή που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης, καθιστώντας τες εύκολες στη χρήση και από άτομα που δεν είναι ειδικοί. Ιδίω μιλώ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Ενώ επίση ο κανονισμό αποκρίνεται και στι ανάγκε όπω οι ηλεκτρονικέ φραγίδε, ηλεκτρονικά τιμολόγια, πιστοποίημα, ηλεκτρονική παράδοση γράφων κτλ. Θα εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία που έχει ξεκινήσει να εμφανίζεται σε διάφορα κράτη-μέλη. Παράδειγμα χάρη σε ό,τι αφορά τη χρονοσφραγίδα, που ξέρουμε ότι η νομοθεσία δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι συνομοθέτες επίσης καλούνται να θεωρήσουν προτεραιότητα την ε, συγκεκριμένη πρόταση και να έχει εγκριθεί μέχρι το τέλος της ε, παρούσας ε, κοινοβουλευτική περίοδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή και τώρα η συνάδελφος Ούλφκοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκόπο έχει να ανοίξει το δρόμο για το δυναμικό που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες ε, στο πλαίσιο ενός ασφαλούς περιβάλλοντος με περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές, διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και, διαχει... και διασυνοριακές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο τις επιχειρήσεις, κυρίως τους ανθρώπους, τους πολίτες. Συνδυάζει την περαιτέρω διάδοση του προγράμματος δράσης ε, της ψηφιακής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την απλούστευση και την ε, ιδιότητα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας σε μια περισσότερο συμμετοχική κοινωνία. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και οι υπηρεσίε εμπιστοσύνη είναι καθοριστική σημασία για όλου, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ και να προστατεύεται η ιδιωτικότητα, ε, ο ιδιωτικό βίο. Αυτό νομίζω ότι θα μα απασχολήσει πολύ και στο μέλλον. Στο έργο του Κοινοβουλίου, ε, καθώ επεξεργαστήκαμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρειαστεί να έχουμε ευρεία αλλά και σταθερή συνεργασία, γιατί υπάρχουν πολλέ τεχνικέ και πολιτικέ πτυχέ που θα πρέπει να αποτιμηθούν, να τι μελετήσουμε. Όπως για παράδειγμα, μόλις ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μία ταυτοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών εθνικών συστημάτων ταυτοποίησης. Θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις, πολλές συζητήσεις για τις επιπτώσεις από την σκοπιά του κόστους, γι' αυτό είμαι ήδη βέβαιη, και για τα επίπεδα της ασφάλειας ή τα όρια της δυνατότητας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, τα κίνητρα που θα δοθούν στα κράτη-μέλη θα συζητηθούν πολύ, ώστε να κοινοποιούν τα συστήματά τους της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Και το θέμα είναι κατά πόσον τα κίνητρα αυτά θα είναι ισχυρά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευέλικτο και τεχνολογικό σουδέτερο νομικό εργαλείο, ώστε να υπάρχει νομική βεβαιότητα και ασφάλεια σε έναν τομέα όπου υπάρχουν απρόβλεπτες τεχνολογικές εξελίξεις κατά κύριο λόγο. Υπ' αυτήν την έννοια η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προσφέρει ένα σύνολο ελαχίστων, ε, εξελαχίστων κανόνων, ε, πράγμα λογικό. Όμω, ε, σκέφτεται και τι κατεξουσιοδότηση πράξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω το κατάλληλο μέσο για να διασφαλίσουμε την ευελιξία. Αυτό το μέρος τη όλη διαδικασία θα απασχολήσει και τις συζητήσει του Κοινοβουλίου καθώς και τη δική μας την εξέταση του θέματος. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό για μας στο Κοινοβούλιο θα είναι το εξή. Να ακολουθήσουμε μία συνολική σφαιρική δυνατόν προσέγγιση για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Οι κανόνες και οι κανονισμοί που θα σχεδιαστούν και θα εγκριθούν θα έχουν επιπτώσεις στους πολίτες και τις αγορές. Γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις είναι αγοριές και ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης διαφορετικών μερίδων του πληθυσμού, διαφορετικών γενεών. Έτσι λοιπόν, να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην ξεχνάμε τι υποκρύπτεται πέρα από τα στοιχεία που, που μελετούμε σε μια πρώτη φάση. Τα ηλεκτρονικά συστήματα, η ηλεκτρονική κοινωνία δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη που έχουν τα αναλογικά συστήματα μεταξύ των πολιτών. Ε, εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι απλώς η τεχνολογία. Είναι το πώς θα οικοδομήσουμε τις κοινωνίες μας σε μια νέα εποχή. Θα ακούσω προσεκτικά τις απόψεις όλων των συναδέλφων για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόσφατα στην έκθεση για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενία αγοράς μιλήσαμε για τα υφιστάμενα κολλήματα όπου ένα από τα θέματα ήταν η εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η προκείμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση τη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να επιτρέψει έτσι ένα ακόμη βήμα, αποτελέσει μάλλον ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Η σχετική οδηγία ίσως προπορεύεται της εποχής της. Συμβαίνει καμιά φορά αυτό με την ομοθεσία. Οι στόχοι της οδηγίας της προδεκαετίας εξακολουθούν να είναι σημαντικοί σήμερα. Δυστυχώς διαπιστώνουμε σήμερα ότι η οδηγία επέτρεψε στις χώρες μέλη να διαθέτουν υπερβολικά ευρύ περιθώριο λιγμών και τελικά γίνεται δύσκολο να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση. Πρόσφατα, στα πλαίσια των δημοσίων προμηθειών, συζητήσαμε και την ψηφιακή διαδικασία ανάθεσης ή δημοσίων προμηθειών. Θα ήταν μεγάλο το βήμα της πρόοδου αν μπορούσαμε να επιτύχουμε να εφαρμοστεί γρήγορα, ταχαίως στην Ευρώπη η ηλεκτρονική ανάθεση. Αυτό θα μπορέσει να γίνει όμως μόνο εφόσον οι προσφέροντες μπορούν να ταυτοποιούνται με τρόπο ελέγξιμο, κάτι το οποίο μέχρι τώρα προκαλούσε προβλήματα νομίζω ότι με το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Επειδή ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή της συζητήσεω, θα περιοριστώ σε λίγα μόνο ουσιαστικά σημεία. Όπως ήδη λέχθηκε, θεωρώ σημαντικό να υπάρξει ευρεία αποδοχή για να υπάρξει και η απαραίτητη εμπιστοσύνη ή ανάποδα. Εδώ τίθεται το θέμα εάν θα πρέπει ίσως ανεξάρτητοι οργανισμοί να ελέγχουν τα συστήματα. Διότι τα περιθώρια λιμών των χωρών μελών δεν έχουν οδηγήσει σε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Απλώς να πει μια χώρα ότι διαθέτω ένα σύστημα και το κοινοποιώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκεί. Χρειάζεται ειδική κοινοποίηση, α το πω έτσι. Με ενδιαφέρει επίση η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και πώ θα εξασφαλιστεί στην πράξη. Διότι αυτή τη στιγμή σκηνοποιηθεί ένα σύστημα πρέπει επίση να εγκριθεί. Επειδή όμω διαφέρουν πολύ τα συστήματα ταυτοποίηση, θα χρειαστεί οι εθνικέ αρχέ να προσαρμόσουν τα συστήματά του ή θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε γενικέ διατάξει που να ισχύουν για όλα τα συστήματα ταυτοποίησης. Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα, αυτό θα χρειαστεί νομική πράξη της Κομισιόν. Έρχομαι σε ένα άλλο σημείο, διότι ο κανονισμός προσφέρει και πολλές βάσεις εξουσιοδότησης της Κομισιόν. Πρέπει να συζητήσουμε αν όλα αυτά είναι απαραίτητα ή αν ορισμένα πρέπει να ρυθμιστούν από τον ίδιο τον νομοθέτη. Γνωρίζω ότι αυτό το, εκεί το πεδίο είναι περιορισμένο αλλά πρέπει να μείνει ανοιχτό και να ηγητηθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Επανέρχομαι στην σημασία των υπηρεσιών αυτών για τους πολίτες. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό περιορισμού της γραφειοκρατίας καθώς και του σχετικού κόστους των συναλλαγών εφόσον προσφέρονται ψηφιακέ υπηρεσίες. Βέβαια, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει ή επίση την λήψη αποφάσεων για τις επενδύσεις στο μέλλον, που δεν πρέπει να επηρεαστούν αρνητικά. Εγώ θεωρώ ότι σωστό είναι να ισχύσει ένας κανόνας ελάχιστων προδιαγραφών για να τηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα και τα στοιχεία κόστους. Να ανασταλούν δε, δε, οι αποφάσεις για επενδύσεις μέχρι να λάβουν τελική μορφή οι αποφάσεις αυτές. Και γι' αυτό απευθύνω έκκληση προς όλους να δράσουμε όλοι ταχαίως. Υπάρχει ακόμα ανάγκη συζητήσεω. ωστόσο χαίρομαι για την ε, πρόταση τη Κομισιόν και θεωρώ ότι προσφέρει επαρκή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστούμε. Ο Νεκότερ. Um, the proposal before us... Ευχαριστώ, Πρόεδρε η πρόταση που έχουμε μπροστά μα μπορεί να αλλάξει πολύ την ψηφιακή οργάνωση τη Ευρώπη ή να έχει διαφορετικό αντίκτυπο από ό,τι νομίζουμε τώρα. Ήταν δύσκολο να ε, υλοποιηθεί η προηγούμενη οδηγία, ίσω να ήταν και υπερβολικά ευέλικτη. Τώρα έχει προσθέσει στην πρόταση Επιτροπή και τι υπηρεσίε εμπιστοσύνη. Αλλά ακόμη και όταν ασχολούμαστε με κάποιο, κάποια σύνολα τη εμπιστευτικότητα ε, τη επιγραμμική, η ταυτοποίηση του ε, προσώπου του καθενό είναι θέμα του ιδιωτικού βίου. Ανέγεται σε αυτή τη σφαίρα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών και σε αυτό το σώμα θέλουμε βεβαίω η υπεράσπιση των δικαιωμάτων να είναι ισχυρή ε, και είναι δικαίωμα των πολιτών μα. Η, η, η τωρινή πρόταση ουσιαστικά θέλει να εξασφαλίσει την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών, όμω κάποιε τεχνολογικές λύσεις θα διασφαλίζουν περισσότερο τον ιδιωτικό βίο και θα ε, κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών περισσότερο από ό,τι άλλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει τα κράτη-μέλη να μην επιβάλλουν συγκεκριμένε τεχνικέ προδιαγραφέ για όσου ε, λειτουργούν και έχουν την έδρα του εκτό τη επικράτειά του, όμω πώς θα εξελιχθούν οι τεχνολογίες που ασχολούνται με την προστασία του ιδιωτικού βίου τη εμπιστευτικότητα. Αυτό είναι ένα θέμα. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή καλό θα να γνωρίζει όλες να αφήσει τις τεχνολογικέ ε, διευκρινήσει κατά μέρο, διότι θέλουμε να υπάρξει συνοχή στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπογραφών αλλά και με άλλες πολιτικές όπως ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Από τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνών ε, που έχουν ε, διεξαχθεί εδώ και χρόνια έχουμε δει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι αρκετά επιφυλακτικοί για το κατά πόσο οι πολιτικοί θύνοντες είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ε, που να τους ικανοποιεί σε σχέση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων τους Οπότε να σκεφτούμε πολύ καλά τι ανησυχίε μπορεί να προκύψουν ω προ την προστασία των δεδομένων. Αυτό ισχύει για τι υπηρεσίε εμπιστοσύνη και του παροχή του, καθώ και την μεταφορά δεδομένων διασυνοριακώ. Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάναμε και στο παρελθόν πολλέ φορέ. Αλλά στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανόνε που ενθαρρύνουν τη δημιουργία, τη νέων συστημάτων μεταφοράς των δεδομένων διασυνοριακώ. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε τους παροχή υπηρεσιών εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης με τεχνολογικά και διοργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε κατά πρώτον τη δική τους ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που προσφέρουν. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς θα ε, ασχοληθεί με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων όταν ε, κάποιε εταιρείε που προσθέτουν τέτοιε υπηρεσίε βρίσκονται εκτό τη επικρατειά μα και με τι ηλεκτρονικέ επιγραφέ. Τι σκεφτήκατε, ποια ήταν η πρόθεσή σα όταν προσθέσατε τον όρο unambiguous, χωρί αμφισημίες δεν είναι μέρο τη κλασική ε, ορολογία που χρησιμοποιείται για να συζητήσουμε την συνολική διαχείριση δεδομένων και τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ. Μιλούμε για τη συλλογή, για την επαλήθευση περισσότερων δεδομένων σε σχέση με ιδιώτε. Μήπω είναι υπερβολική συγκέντρωση δεδομένων. Εδώ να είμαστε προσεκτικοί ω προ τον ιδιωτικό βίο και την εμπιστευτικότητα, λόγω χάρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τσεκάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, έχουμε διερμηνία από τα ρουμανικά. Mm-hmm. Ωραία. Θα μιλήσω λοιπόν ρουμανικά. Κατά πρώτον, ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευκαιρία που μας δίνει να συζητήσουμε το θέμα αυτό με αφορμή τη σύντομη παρουσίασή της. Ίσως χρειαζόταν μια περισσότερο τεχνική αναδρομή, διότι η οδηγία αυτή και η πρόταση κανονισμού είναι από τους πρωταρχικούς στόχους που είχε αναλάβει στη φάση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την ψηφιακή της ατζέντα. Εάν θέλουμε να υπάρξει εσωτερική αγορά στον ε, τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, σίγουρα χρειάζεται διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η ισχύουσα οδηγία υλοποιήθηκε με τρόπο κατακαιρματισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή διαφορετικά από το ένα κάτω μέλο στο άλλο. Το γεγονό αυτό οδήγησε σε έλλειψη διαλειτουργικότητα. Ακούστηκε και ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η χρήση ηλεκτρονικών καρτών ταυτοποίηση σε πολλά κράτη-μέλη. Δυστυχώς, σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε μόνο μερική διαλειτουργικότητα. Έχει εκπονήσει αρκετέ μελέτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου έχει καταλήξει ότι όντω τα συστήματα ηλεκτρονική διαχείριση υπάρχει περιορισμένη και μερική διαλειτουργικότητα. Αυτό δείχνει ότι η οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές προφανώς ε, υλοποιήθηκε μόνο μερικώς. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να ε, ταυτοποιηθεί κανείς στο πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρονικής ε, διαχείρισης. Κάποια συστήματα είναι πολύ απλά με τη χρήση κωδικού και password κωδικού πρόσφασης, κάποια άλλα είναι ιδιαίτερα προηγμένα. Για την ίδια υπηρεσία δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων ταυτοποίησης στις διαφορετικές χώρες. Άρα έλλειψη λειτουργικότητας και εδώ. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι οι πιστοποιημένες, μάλλον οι παροχές υπηρεσιών πιστοποίησης μπορεί να έχουν λάβει και να μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα, άδεια και να μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα μέλο. αλλά να μην έχουν το απαιτούμενο επίπεδο ε, αξιοπιστίας και έγκριση ώστε να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες χώρες. Μπορεί να είναι δηλαδή εθνική η έγκρισή τους. Εδώ λοιπόν είμαι ιδιαίτερα περίεργη αν έχετε κάτι να πείτε για κάτι σαν ηλεκτρονική γέφυρα, μια πασαρέλα που να διασυνδέει τα συστήματα αυτά μεταξύ τους. Όλα αυτά έχουν ε, στενή σχέση και με την ε, οδηγία για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, την τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και το καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι έχει κάνει ήδη ένα σημαντικό βήμα. Το 2009 ή 10, αν καλά, όταν ενέκρινε νομοθεσία για τις υπηρεσίες ταυτοποίησης. Στηρίζω αυτά που είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι, διότι δεν αρκεί να έχουμε απλώς ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα. Μιλάμε για μια αγορά παγκόσμια πλέον. Θέλουμε να έχει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε τη διαλειτουργικότητα με παρόμοιες υπηρεσίες που προέρχονται ενδεχομένω από τρίτες χώρες θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πετύχουμε το ένα επαρκέ επίπεδο διαλειτουργικότητα για το σκοπό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν, εάν έχετε κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε, κυρία Τσικάου. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, um, thank uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε και κύριοι βουλευτές για τις αρχικές σας αντιδράσεις. Εδώ θέλουμε να έχουμε στενή συνεργασία στο ερχόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να εξεύρουμε και τις κατάλληλες λύσεις για ένα ζήτημα τόσο σοβαρό. Ήθελα να αναφερθώ στη μελέτη τύπου που ετοιμάσαμε κατά την προετοιμασία επίσης της πρόταση του κανονισμού εδώ. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τις διαφορετικές επιλογές και αξιοποιήσαμε και το πολύτιμο έργο του Κοινοβουλίου από το παρελθόν. Είδαμε τι μπορεί να γίνει με μια, μια εργαλειοθήκη, νομοθετική εργαλειοθήκη όπως ε, λέγεται και την υλοποίησή της και μια από τις προτάσεις που εσείς ρίξετε στο τραπέζι σήμερα είναι το αν θα... γιατί υπάρχει πρόταση για εθνικά υποπτικά συστήματα αντί για κάτι που να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη μελέτη δικτύπου αναλύσαμε το κατά πόσον είναι εφικτό το ένα ή το άλλο σύστημα, το εθνικό ή το ευρωπαϊκό ως προς την αποτελεσματικότητα. Αλλά και ανάλογα με το κατά πόσον είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο από τα κράτη-μέλη. Είναι αυτονόητο ότι κάτι που θα γινόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν ε, ιδιαίτερος αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο, αλλά ως προς το κόστος συμπεριλάβαμε κάποιες πληροφορίες και στη μελέτη αντικτύπου και συγκρίναμε το κόστος για τις δύο διαφορετικές επιλογές, οπότε ήταν κάπως παρόμοιο. Το ευρωπαϊκό επαπτικό σύστημα δεν θα συνείδε πλήρως με την αρχή της επικουρικότητας. Γι' αυτό προσπαθούμε να... Γι' αυτό έχουμε κάνει τις συγκεκριμένες προτάσεις στο σχέδιο κανονισμού. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επηρεάσει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και να την ρυθμίσει. Αυτό το προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι κάτι που ε, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συμφωνώ με κάτι που υπόθηκε σήμερα, ότι ένα από τα καθοριστικά σημεία για την επιτυχή υλοποίηση θα είναι να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία και να καλύψουμε τα ζητήματα της προστασίας των δεδομένων. Συμφωνώ απολύτως με κάτι άλλο που επίσης ακούστηκε, την συζήτησή μα εδώ, ότι πρέπει να δούμε πώς θα προασπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό είναι και κάτι άλλο που ακούσαμε σήμερα, ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από την πείρα μας της κακής υλοποίησης της οδηγίας του 1999. Ένα σημαντικό στοιχείο που το αναφέρατε κι εσείς ξανά και ξανά στη συζήτηση είναι η διαλειτουργικότητα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τέτοιες λύσεις που στο, διαρκώ, στο ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον να είναι και ικανοποιητικές. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στενά ώστε οι δύο συνομοθέτες να προχωρήσουμε σταθερά στον δρόμο αυτό. Ο κανονισμός αυτός είναι ένα καθοριστικό ε, στοιχείο στην οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς, αλλά πρέπει να βρούμε και τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις. Θέλουμε αυτή τη φορά να λειτουργήσει αυτή η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό θα συνεργαστούμε στενά με τους εισηγητές σας και ελπίζουμε οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ικανοποιήσουν τι ανάγκε των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Για να κλείσουμε, να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μα, κυρία Ουλφκοκ. Εάν θέλετε, έχετε το λόγο. Ε, well, thank you. Ευχαριστώ. Νομίζω αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων πριν γυρίσουμε στις πατρίδες μας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά δείχνει ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα. Είναι τεχνικό. Και αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάποιο βαθμό. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, για ζητήματα της αγοράς και καταλήξαμε στην ουσία, στην ουσία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μάλλον καλό, γιατί εάν το διατηρήσουμε αυτό στο νου μας και δεν παγιδευτούμε στις λεπτομέρειες, παρόλο που και αυτές θα να τις φροντίσουμε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θέλουμε λύσεις καλές με χαρακτήρα σφαιρικό. Να μην καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που είχαμε με την προηγούμενη οδηγία. Ήταν αρκετά περιττή και μάλλον χάσιμο χρόνο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας για τις συνεισφορές σας και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κυρία Ολφκοκ. Να θυμίσω ότι η εξέταση του Σχεδίο έκθεσης ε, προβλέπεται για τις 18-19 Μαρτίου του 2013 και τότε θα ξανακούσουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ ε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσέλευσή του και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Παρουσίαση από την Επιτροπή της ανακοίνωσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις ευθύς πόλεις και κοινότητες. μαζί μας έχουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κύριο Τάτσινέσκου Thank you, President. Thank you, uh, members of uh, this committee. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα την ανακοίνωση για τις ευφύς πόλεις και κοινότητες και την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση Καινοτομία εκπροσωπώ μια ομάδα που συγκροτήθηκε εντό τη Κομισιόν. Ε, την Κερκάλα και Κρού είναι οι αρμόδιοι επίτροποι για ενέργεια, μεταφορέ ε, και τεχνολογίε επικοινών πληροφοριών αντίστοιχα και κάποιε άλλε γαμαδέλτα συνεργάζονται. Έχουμε λοιπόν συγκεντρώσει στην τεχνογνωσία μας τη χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσουμε μια πολύπλοκη πρόκληση, δηλαδή τη δημιουργία πιο βιώσιμων πόλεων και κινητών στην Ευρώπη και ελπίζουμε και με τους συμπολίτε, αλλά και με εσά να έχουμε συνεργασία για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ο Μπάν Κιμούν είπε νωρίτερα ότι οι ενεργειακέ κλιματικέ προκλήσει ε, θα τι κερδίσουμε, θα τι χάσουμε στι πόλει. Το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στι πόλει και οι αστικέ μα δραστηριότητε, ε, επιχειρήσει, πολίτε, δημόσιε υπηρεσίε παράγουν το 70% των θερμοκηπιακών αερίων και χρησιμοποιούν το 70% τη ενέργεια. Επομένως θεωρούμε ότι μια από τις μεγαλύτερες δυνατότητες που έχουμε για σύγκληση μεταφοράς ενέργειας τηλεπικοινωνιών και σχετικών υπηρεσιών θα είναι στις πόλεις. Ήδη οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά ε, σε τεχνολογίες εφιών πόλεων. Το Fast Company βάζει την ε, Βιέννη στην πρώτη θέση, της πιο εφιούς δηλαδή πόλεις ε, και 6 στις δέκα είναι ευρωπαϊκές πόλεις. Οι πόλεις έχουν καταφέρει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουν επενδύσει ήδη σε λύσεις για την κινητικότητα, ICT, για μείωση της ε, κατανάλωσης ενέργειας, αλλά δεύτερον έχουν επίσης καταλάβει ότι μία πόλη για να είναι ευφύης δεν θα πρέπει αυτό να συνιστά μια πρόκληση μόνο τεχνική τεχνολογική, είναι διεπιστημονικό ε, θέμα και προμηθευτές, ε, χαράκτες πολιτικής, ακαδημαϊκοί ερευνητές, χρηματοδότες και όλοι ε, άλλοι πρέπει να συνεργαστούν σε πολλά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτή εμπειρία στην πρώτη και εφαρμογή αστικών προγραμμάτων, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στις τεχνολογίες πληροφοριών επικοινωνιών. Μέχρι στιγμή τα σχέδια αυτά δεν έχουν ε, ενταχθεί ε, στους, ε, σε όλους τους τόμεις εκεί που μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και βέβαια αυτό συνιστά μια χαμένη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης καινοτομίας φύης πόλης και, κοινοτο... και κοινότητες ή κοινωνής τον Ιούλιο. Με σημαντικότερο στόχο αυτής της πρωτοβουλίας αυτής εταιρικής σχέσης είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών εφιών πόλεων ε, ταχύτερα σε ευρωπαϊκές πόλεις και κοινωνίες. Και θα είναι ανοιχτή αυτή η εταιρική σχέση γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν πολλοί. Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή, αυτή η προσέγγιση ευρωπαϊκή εταιρική σχέση είναι κατάλληλη για να πετύχουμε του στόχου μα. Οι εταιρικέ σχέσει καινοτομία είναι ένα πλαίσιο που φέρνει κοντά όλους τους εμπλεκομένους φορείς, αναξάρτητους πολιτικής υπηρεσίας, συνόρων για την επιτάχυνση της καινοτομίας, αντιμετώπιση μιας σημαντικής κοινωνικής πρόκλησης για την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και βέβαια η εταίροι είναι το σημαντικό στοιχείο. Η Κομισιόν δεν θα είναι εταίρος, θα είναι όμως ε, ένας ε, υποστηρικτής. Οι ε, δραστηριότητες τώρα αυτής της συγκεκριμένης εταιρική σχέση, θα βασίζονται σε τρία είδη δράσεων που θα τις μελετήσουμε ακόμη πιο διεξοδικά. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ή μια κοινότητα πόλεων, Πέρυσι ξεκινήσαμε τη λεγόμενη Smart City Stakeholder Platform που έχει προσελκύσει πάνω από 6.000 άτομα μέχρι τώρα, άτομα που εργάζονται για δημόσια τομέα, ερευνητικά ιδρύματα, χειρίς και μπορούν να παράσχουν πληροφορίες για το πώς θα προχωρήσουμε. Δεύτερον, οριζόντιες δράσεις για τη δημιουργία πλαισίων για την ανάπτυξη λύσεων ευφυών πόλεων ε, σε βιομηχανικό επίπεδο. Παραδείγματο χάρη, δημιουργία θέσεων στην αγορά για προμηθευτέ και πολιτέ υπηρεσιών προϊόντων, καλύτερη χρήση των ε, δημοσίων προμηθειών, τυποποίηση, ρύθμιση, στήριξη καινοτομία στι τοπικέ ε, αυτοδιοικήσει και τρίτον, βελτίωση τη πρόσβαση και χρήση του δημοσίου τομέα σε άλλε η τρίτη οριζόντια δράση θα είναι η ανάπτυξη και η συγχρηματοδότηση κάποιων σημαντικών ε, εμβληματικών σχεδίων που ενσωματώνουν τεχνολογίες, ε, κινητικότητα, τύπη ε και συνεργασία όλων των επιπέδων, τοπικών, περιφερειακών κτλ. Το σημαντικότερο όμως κομμάτι της εταιρικής σχέσης ουσιαστικά είναι η δημιουργία τοπικών περιφερειακών εταιρικών σχέσεων που θα εκμεταλλεύεται την εμπειρία που συλλέγεται, θα αναπτύσσει λύσεις και έχει και αρκετά πλεονεκτήματα. Για το δημόσιο τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δοκιμασμένες, αποδεδειγμένες λύσεις που όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν στους τοπικούς περιορισμούς, τοπικές συνθήκες. Για τους πολίτες, ε, νέες απλές ε, λύσεις ε, αποδετικές ω προς το κόστος, το ίδιο και για υπηρεσίες, λύσεις διαλειτουργικές και λύσεις βιώσιμες από οικονομικής πλευράς. Για τον ιδιωτικό τομέα τα πλεονεκτήματα είναι ότι θέλουμε να έχουμε θετικές επιχειρηματικές ε, πρακτικές που θα βοηθήσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη όλων των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται διότι βλέπουμε πολλή τεχνολογία αλλά λίγη ανάπτυξη αυτή της τεχνολογίας. Και βέβαια και έχουμε διάφορες δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη, έχουμε τα δίκτυα γεφή πόλη στην Ευρώπη, έχουμε διάφορα, το Civitas, Green Digital Charter και πολλά άλλα. Τέτοια παραδείγματα. Επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε και τη χρηματοδότηση μέσω του ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, Έχουμε πρωτοβουλίε όπω το Green V, καλή κοινοπραξίε ή συμπράξει δημόσιο δικού τομέα. Θέλουμε να κοινοπραξία, Η συμπραξει δημοσιο τομεα θελουμε να στηριξουμε πρωτοβουλία προγραμματισμού Joint Europe και ένα κοινό πρόγραμμα επίσης για τις ευφυείς πόλεις. Και η ΕΤΕΠ θα βοηθήσει στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τελικά έναν αγωγό μέσω του οποίου θα παρέχονται νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και σχετικά ζητήματα. Θα χρησιμοποιήσουμε και τον ορίζοντα 2020 και βέβαια στη συνέχεια θα έχουμε και δράσεις ανάπτυξης με τη μορφή τοπικών εταιρικών σχέσεων και συμπράξεων. κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής ε, Εταιρικής Σχέσης και Ενοτομίας. Σε ευρύτερη κλίμακα από τη σήμερα όλα αυτά. Το πρώτο τμήμα λοιπόν αυτού του αγωγού, αν θέλετε, είναι ορίζον 2020 και εξαρτάται από την διάθεση παρκούς χρηματοδότησης για όλους τους τομείς αυτούς. ΤΠΕ, ενέργεια, μεταφορές. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι για μας είναι προφανές ότι το 20% μείωση τη χρηματοδότηση για τι μεταφορέ στον ορίζοντα 2020 είναι κάτι που μα ανησυχεί και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κάποιε από τι φιλοδοξίε μα και του στόχου μα. Και με άλλες εταιρικέ σχέσεις καινοτομία πάλι πρέπει να μα δώσει το Συμβούλιο το πράσινο φω για να δημιουργήσουμε τη δομή, να ιεραρχήσουμε τι προτεραιότητέ μα, τι ενέργειε μα, να έχουμε και ένα σχέδιο στρατηγική υλοποίηση και να προχωρήσουμε περιμένουμε όλα αυτά να γίνουν επί Ιρλανδικής Προεδρίας, σύντομα δηλαδή, και ελπίζουμε αυτή η συγκεκριμένη εταιρική σχέση καινοτομία να είναι πλήρως επιχειρησιακή μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ήδη την υποστήριξή του για την έννοια Ευρωπαϊκών Εταιρικών Σχέσεων Καινοτομία ήδη από το 2010. Και βέβαια, προφανώ περιμένουμε να συνεργαστούμε μαζί σα και για τη συγκεκριμένη εταιρική σχέση. Και εδώ, κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω την ε, εισαγωγική μου παρουσίαση. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την παρουσίασή της. Ζητά κάποιος ε, συνάδελφος τον λόγο. Κανείς ή καμία. Αποτέλεσε το τελευταίο σημείο συζήτησης για φέτος. Να κλείσουμε λοιπόν και να θυμίσω σε όλους ότι θα ξαναβρεθούμε στις 23 και 24 Ιανουαρίου του χρόνου. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στήριξή της σήμερα και εύχομαι σε όλους καλές γιορτές στο επανειδήμιο.